Doamnă președintă! Ah. <laughs> Good afternoon, colleagues. Χαίρετε, αγαπητοί συνάδελφοι. Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Θα πρέπει να σας ενημερώσω ότι τα χθεσινά συνοπτικά πρακτικά καθώς και τα κείμενα που εγκρίθηκαν